πριν απευθυνθώ και καλωσορίσω τον πρόεδρο της Γουινέας, θέλω να σας πληροφορήσω για αυτό που έγινε στη Λιέγη, στο Βέλγιο. Ένας άντρας δολοφόνησε δύο Βέλγους αστυνομικούς και έναν Βέλγο πολίτη. Στη συνέχεια ε, και ο ίδιος πυροβολήθηκε και έχασε τη ζωή του. Ε, πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Δεν ξέρουμε αν είναι τρομοκρατική επίθεση ή όχι. Όμως βρισκόμαστε στο πλευρό του βασιλείου του Βελγίου, στο πλευρό των πολιτών του Βελγίου και στο πλευρό των οικογενειών των δύο αστυνομικών και του Βέλγου πολίτη που έχασαν τη ζωή του σήμερα το πρωί στη Λιέγη. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο της Γουινέας που μας έστειλε τα συλληπιτήριά του για την επίθεση αυτή. Δεν ξέρουμε αν ε, ήταν τρομοκρατική υπόθεση ή όχι τρομοκρατική επίθεση μάλλον ή όχι, αλλά για άλλη μια φορά στην Ευρώπη και στο Βέλγιο θρυνούμε νεκρούς εξαιτία μιας ε, ακατανόητης βίας. Συνάδελφοι, είναι μεγάλο μου χαρά που μπορώ σήμερα στο ημικυκλευτό να υποδεχτώ τον πρόεδρο της Γουινέας Αλφα Κοντέ. Κύριε Πρόεδρε, είστε ένας Αφρικανός Πρόεδρος που έρχεται να απευθυνθεί στην Ολομελιά μας. Η συνάντηση αυτή